το οποίο σήμερα Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απόψε όπως βλέπετε το κάναμε ένα μεγάλο στούντιο, στούντιο τηλεόρασης. Σήμερα συμβρισκόμαστε σε αυτή την ε, ημερίδα, σε αυτή τη μέρα εκλογών που όλοι οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν το ποιο από του υποψηφίου θα λάβει έδρα εδώ, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συζητήσουμε τώρα για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μιλήσουμε σε διαφορετικέ γλώσσε. Έτσι είναι η Ευρώπη. Είμαστε εδώ, κόσμος από όλες τις χώρες, από διαφορετικές ε, κουλτούρες, χάρη στη σκληρή δουλειά των ε, διερμηνέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε επομένω έτσι να συνεννοηθούμε και θα συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό, αυτό είναι η συζήτησή μας. Κβο Vadis Europe. Πού πας Ευρώπη. Θα συζητήσουμε επομένω εδώ πέρα με την Κομισιόν, με το Κοινοβούλιο, τι θα γίνει με τη συνθήκη τη Ευρώπη, τι θα γίνει με τη συνθήκη τη Λισαβόνα επομένω, πώ θα γίνει με την κρίση, θα γίνει με του και να δούμε ποιοι θα είναι μαζί μα για αυτή τη συζήτηση πρώτα-πρώτα. Έχουμε την Μάργκοτ Βάλστρομ. Προέρχεται από την Σουηδία και είναι αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Είναι η επίτροπο, η οποία έχει το χαρτοφυλάκιο των θεσμικών ζητημάτων και στατική επικοινωνία, τόσο ώστε να μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει στου Ευρωπαίους τι είναι η Ευρώπη, Πώ δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλησπέρα σα κυρία. Καλησπέρα λέει κύριε Βάλστρομ και στη συνέχεια ο Μάριο Σέπη είναι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού και Κοινωνικού Συμβουλίου. Είναι Ιταλός, έχει βαθιά γνώση των κοινωνικών θεμάτων και δικαιωμάτων, αλλά επίση ξέρει και την σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Καλησπέρα, λέει ο κύριο Σέπε. Κατά τρίτον, άλλο Ιταλός, Ρικάρντο Πέρσιτ είναι μέλο του ιδρύματο Εξωτερικών Υποθέσεων και επίση έχει μια μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την οικονομία και τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Καλησπέρα και σε εσά. Αλλά θα πρέπει να υποδεχτούμε και τον Χωσέ Μαρία Κασάτο που είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Κόρδοβα και κατέχει την έδρα Ζα Μονέ για θέματα ευρωπαϊκά και οικονομικά και επίσης ξέρει τα θέματα της ε, νομισματικής ένωσης. Καλησπέρα και σε εσά, αλλά έχουμε και τον Ρίτσαρντ Σίνοτ, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου. Είναι ειδικό στα θέματα κοινή γνώμη. Και επίσης ε, ξέρετε τα του Ευρωμαρόμετρου, ξέρετε τα της πολιτικής στην Ευρώπη. Γεια σας και σας και επίσης έχουμε την Χριστίνα Σιγανίδου, δημοσιογράφος, Ελληνίδα, της ΕΡΤ 3. Καλησπέρα Χριστίνα. Τώρα πώς να πω το όνομα της Ντομινίκας που είναι εδώ, λέει Ντομινίκα Ψετσολκόφσκα. Ε, εργάζεται για την εφημερίδα Γκαζέτα Βιμπόρσκα, ε, μία από τις πιο έγκυρες της Πολωνίας αλλά και τις πιο έγκυρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Comenzamos eh, existen eh, Ένα από του προβληματισμού ενισχύει για τι εκλογέ είναι το θέμα τη συμμετοχή τη αποχή. Δεν ξέρω οι εντυπώσει σα πώ έχουν μέχρι στιγμή για την αποχή, για το πώ κόσμο κατέβηκε στι εκλογέ. Ανάμεικτε είναι οι εντυπώσει. Έχουμε 4-5 χώρε όπου μάλλον αυξήθηκε η συμμετοχή. Αλλά στις υπόλοιπες, στις περισσότερες χώρες μέλη τα πράγματα είναι τα ίδια. Μία από τα ίδια όπως και τις τελευταίες εκλογές. Στις ορισμένες χώρες μέλη έχουμε ακόμα λιγότερη συμμετοχή και βέβαια έχουμε κάποιους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό και από ό,τι φαίνεται από τις στατιστικές του βαρόμετρου είναι η εσωτερική πολιτική. Τι γίνεται στο εσωτερικό κάθε κράτος μέλους, πόσο μπαίνει η Ευρώπη στο, στο πολιτικό προβληματισμό και ε, αυτό διαμορφώνει το πώς βλέπουν τις ευρωεκλογέ οι ε, πολίτες και να το ασκούν το δικαίωμα του να ψηφίσουν. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, άπαξ και ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει περισσότερη εξουσία γιατί κατά τον τρόπο θα έχει πιο συρρυκνωμένη εκπροσώπηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω, κύριε Βαλστρομ, και θέλουμε όσο γίνεται περισσότερη συμμετοχή, έτσι θα αυξηθεί η νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωβουλευτών καθέκαστον. Ακριβώ όπω θα ίσχυε και για ένα εθνικό κοινοβούλιο. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κατόφλι για την νομιμότητα, γιατί η δημοκρατία δεν είναι κάτι το στατικό. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, μεταβάλλεται. Επομένως θα πει είναι ένας συνεχής ε, αγώνας, διαδικασία. Κάτι το οποίο ξεκινά για φετήρια, ρίζες στην εσωτερική εθνική πολιτική και κουλτούρα. Όπου πολλές φορές τα πρόσωπα μετράνε περισσότερα εδώ από τις εθνικές εκλογές και ο κόσμος διαλέγει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τις εκλογές. Όμως είπατε τη λέξη ευρωβαρόμετρο, οπότε πάμε στον κύριο Σύνοδο. Τι λέτε εσείς που ζητείτε το λόγο. Πάρα πολύ σημαντικό το να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε όλο ένα και πιο ευξημένη συμμετοχή. η Δανία και άλλες δύο χώρες έχουν αυξημένη συμμετοχή όπου στην, ε, στη Δανία ξέρουμε ότι θα έχουμε δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Η προσπάθεια που γίνεται μέσω του δημοψηφίσματος αυτού είναι να μην ε, περιορίζεται η διαδοχή του χρόνου μόνο στους άρενες εκεί έχει υπάρξει μια μικρή πτώση. Και υπάρχουν κάποιες χώρες επίσης στις οποίες η συμμετοχή παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα. Δεν έχουν υπάρξει κάποιες ριζικές αλλαγές. Έχουμε, Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το, την ηχοληψία όσον αφορά τον κύριο Σύνος που δεν ακούγονταν καθόλου καλά. Είπαμε ότι συνοούμαστε, μεταφραζόμαστε, αλλά πρέπει να δουλεύει και το μικρόφωνο. Θέλετε να τα πω από την αρχή. Ναι, ναι, ναι, φοβάμαι, ναι. Πολύ καλά. Καλώς λοιπόν. Ποια είναι η ερώτηση καταρχάς. Εσείς μας μιλήσατε για το Ευρωβαρόμετρο και για τα προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί τελευταία. Θα συμφωνήσω με την Επίτροπο Βάλστρομ για τη σημασία που έχει η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Είναι κάτω του 50%. 45 με 50% ανάλογα πώς το μετράει κανείς. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αν θέλει κανείς να απεικονίσει τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα διάγραμμα, θα δει ότι ανεβαίνει συνεχώς. Ενώ ταυτόχρονα από το 1979 η συμμετοχή στις εκλογές είναι ένα γράφημα το οποίο κατεβαίνει συνεχώς. Και αυτό είναι συνεχές σαν φαινόμενο. Συνεπώς βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση σήμερα ε, με αυτήν που διαπιστώσαμε στις ψηφοφορίες που έγιναν στα μέσα της εβδομάδας. Σε τρεις χώρες υπήρξε άνοδος στη συμμετοχή. Στην Δανία τελικά υπήρξε άνοδος, είναι σαφές. Γιατί ξέρετε ότι έγινε και δημοψήφισμα για τις διακρίσεις ε, στο φύλλο του διαδόχου ε, για τον θρόνο στην χώρα, δηλαδή να μην περιορίζεται μόνο σε ε, άρενες ή να μην διευκολύνονται περισσότερο οι άρενες διάδοχοι. Εν πάση περιπτώσει τα προβλήματα είναι δεδομένα. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να αντιστοιχίσει τις προεκλογικές διαδικασίες με τα πεπραγμένα και με τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί είναι χαμηλή η συμμετοχή. Δύο παράγοντες νομίζω ίσως να εξηγούν. Καταρχάς, είναι εθελοντική η συμμετοχή στις εκλογές και τελικά ίσως να μην είναι η καλή ιδέα να γίνεται η διαδικασία αυτή η εκλογική ένα τόσο ωραίο ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο στις περισσότερες χώρες. Ίσως θα ήταν προτιμότερο πρακτικά να γίνεται στα μέσα της εβδομάδας όταν ο κόσμος ασχολείται με τα επαγγέλματά του, με τα σχολεία κτλ. Αυτό είναι όμως ένα πρακτικό σημείο θα έλεγα. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές απορίες για να εξηγήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Βέλγιο δεν είδαμε να υπάρχει πάρα πολύ ήλιος. Βέβαια στην Ισπανία ήταν ηλιόλουστη ημέρα. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει η μέρα διεξαγωγής των εκλογών. Να μην συμπίπτει ας πούμε με διακοπές. Ε, δύσκολο είναι αυτό να προγραμματιστεί μακροπρόθεσμα και μάλιστα ε, συγκεκριμένη εποχή. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Το βασικό στοιχείο είναι ότι ε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαδικασία αυτή που ξεκίνησε το 1979 και συνεχίστηκε μέχρι το 2004 και σήμερα ε, με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν νομίζω θα πρέπει να μας αποθαρρύνει σε καμία περίπτωση για το μέλλον της Ευρώπης και το πώς θα σκεφτούμε και τι προσδοκίες, τι όνειρα θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, αυτό που θα πρέπει να ενισχύσουμε είναι η εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση για την Ευρώπη. Να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στον κόσμο. Διδάσκεται και η Ευρώπη όπως τα πάντα διδάσκονται. Μπορείς να φέρεις πιο κοντά τον πολίτη στην Ευρώπη μαθαίνοντάς του και καθιστώντας τον υπεύθυνο. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα και εν ώψη τη Σύνδεξη Λισαβόνα που θα ενισχύσει πάρα πολύ, όπω γνωρίζουμε, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσμικό παιχνίδι τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτές τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους ε, και τις εξουσίες τα θεσμικά όργανα. Θα είναι τεράστια σημασία στο μέλλον αυτό. Κύριε Σέπη, αν είχαμε θεσμικά όργανα ευρωπαϊκά πιο ισχυρά ενδεχομένως με περισσότερες εξουσίες να το αντιλαμβανόταν αυτό ο Ευρωπαίος πολίτης και να τη θεωρούσε πιο κοντά του τα όργανα αυτά. Η αίσθησή μου είναι ότι τα προβλήματα δεν είναι επιμελητιακού χαρακτήρα, δεν είναι πρακτικά, δηλαδή δεν εξαρτάται η συμμετοχή από τη μέρα που θα γίνονται οι εκλογές. Τα προβλήματα είναι βαθύτατα πολιτικά. Και εγώ δεν πήγα να ψηφίσω και ε, αναρωτήθηκα γιατί έπρεπε να ψηφίσω, γιατί δεν έπρεπε να ψηφίσω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν πολλά εμπόδια. Ένα εμπόδιο είναι οι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσει συστηματικά υπονομεύουν την Ευρώπη. Και κάθε φορά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα λένε ότι φταίει η Ευρώπη και όχι οι δικέ του ανεπάρκειε. Δεύτερος, εμπόδιο. Η προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ δεν είχε καμία σχέση με την Ευρώπη. 27 εθνικές αυστηρά προεκλογικές εκστρατείες. Καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Μόνο για τα εθνικά προβλήματα της κάθε χώρας. Εμείς κάναμε σαν Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μια μικρή έρευνα και είδαμε ότι σε πάνω από 20 χώρες, 20 από τις 27, η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά τον συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο πώς να ενδιαφερθεί κανείς για την Ευρώπη. Και φυσικά στη χώρα σαν τη δική μου την Ιταλία έγινε μια προεκλογική εκστρατεία εντελώς διαφορετική, ιδιόρυθμη θα έλεγα, και στο ε, Βέλγιο η προεκλογική εκστρατεία αφορούσε περιφερειακά προβλήματα, εθνοτικά προβλήματα και σε άλλες χώρες όπως η Ολλανδία υπήρχαν θέματα φορολογικά κτλ. Αυτό ήταν το δεύτερο εμπόδιο, το τρίτο εμπόδιο. Παρόλες τις προσπάθειες της Μάρκο Φάλστρον η ευρωπαϊκή εικόνα είναι μια εικόνα μακρινή και γραφειοκρατική για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό προκαλείται ε, από το ότι ποτέ δεν προσπαθούμε να φτάσουμε συναισθηματικά στον Ευρωπαίο πολίτη. Εγώ θυμίζω ότι η Ευρώπη έχει μια μεγάλη αποστολή να δημιουργήσει κοινωνική πρόοδο και να καθοδηγήσει την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με κοινωνικούς κανόνες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ο κόσμος δεν θα ενδιαφέρεται και δεν θα πηγαίνει να ψηφίζει. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι απεσιόδοξος τα αποτελέσματα είναι πάνω κάτω σε επίπεδο συμμετοχής τα ίδια με τις προηγούμενες ευρωεκλογέ. Και θυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομιμοποιείται σαφέστατα μέσω των προτάσεών του για το πώ θα βγει η Ευρώπη από την κρίση. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τις σωστές κατευθύνσεις μετά την υιοθέτηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα με περισσότερε ε, αρμοδιότητες σε επίπεδο συναπόφαση, τότε θα ενδιαφερθεί ο κόσμο πολύ περισσότερο. Ήρθε η ώρα. Είναι 9. Οπότε τώρα θα έχουμε την συμμετοχή της ΕΡΤ3. Χριστίνα, είναι δική σου σειρά να πάρεις τη σκητάλη. Κύριε Σύνοτ, τι θεωρείτε, η υπόθεση συνθήκης Λισαβόνας θα έχει happy end. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, γιατί ακόμα ε, δεν, δεν, δεν μεταφράστηκε αυτό το οποίο είπατε. Θεωρείτε ότι η διαδρομή ε, της συνθήκης της Λισαβόνας θα έχει αίσια κατάληξη. Σύνοτ. Όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα καταδεικνύουν στο, στην καταφατική απάντηση, διότι θα ε, έχουμε στη συνέχεια ένα 60% και πάνω επίπεδο ε, συμφωνίας, σύμφωνης γνώμης. Ε, έχουμε και δείγμα του Φεβρουαρίου της Ιρλανδίας, έχουμε τις επαφές οι οποίες έχουν κριθεί επιτυχής μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο. Τον Ιούνιο θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή, πάρα πολύ σημαντική. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε και το θέμα το ότι όταν επαναλαμβάνεται το δημοψήφισμα τότε το καλοσκέφτεται ο ψηφοφόρος, ε, οριμάζει κατά κάποιο τρόπο. Ε, γίνονται και κάποιες εκστρατείες ε, και αλλάζουν οι απόψεις. Σκεφτείτε όμως και το πει τι έγινε στη Βρετανία. Ναι, λέει η κυρία Σιγανίδου. Ας πούμε ότι οι Ιρλανδοί λένε ναι, οι Τσέχοι προσυπογράφουν την συνθήκη και τελικά ο Ντέιβιτ Κάμερον κάνει αυτό το τόσο αγαπητό το δημοψήφισμα. Εξαρτάται από τις συνέπειες, λέει ο κύριο Σινότ. Εάν εξαρτάται από, από τη σειρά των γεγονότων, ούτως ώστε έτσι όπως το είπατε δεν θα υπάρξει πρόβλημα μια που οι Βρετανοί θα πρέπει να κρίνουν από μόνοι τους το τι θα κάνουν. Αν έχουμε όμως μια αλλαγή στην κυβέρνηση ε, και με τον ε, κύριο Κάμερον στα Ινία τότε θα προχωρήσει στο δημοψήφισμα πριν ψηφίσουν οι Ιρλανδοί, οπότε τα πράγματα θα είναι σοβαρά, γιατί θα πούνε οι Ιρλανδοί, ε, ναι, αλλά για κοιτάξτε τι κάνανε οι Βρετανοί, δεν είναι δική μας πια η ευθύνη, να περιμένουμε τι θα κάνουν οι Βρετανοί, οπότε Μπορεί να οι Ιρλανδοί, να, δεν το κάνανε οι Άγγλοι, το κάνουμε εμείς ε, και τελικά να προχωρήσουν στο ναι. Ερώτημα προ την κυρία Βάλστρομ. Τι λέτε όσον αφορά την εκλογή του νέου Προέδρου του... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρείται να γίνει αυτό μετά το δημοψήφισμα όπω προτείνει και ο Σαρκοζή Βάλστρομ. Νομίζω ότι από αυτού θα πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν τον Ιούνιο στο Συμβούλιο οι Κρατών και Κυβερνήσεων. Σε αυτού απόκειται να αποφασίσουν όσον αφορά την ακολουθία, τη σειρά κατά την οποία θα λάβουν χώρα αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε κάποια πρόγνωση. Κύριε Κασάδο, τι λέτε, οι σοσιαλιστές θα έπρεπε να κατεβάσουν δικό τους υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κασάδο, δεν είμαι ειδικό ε, στην πολιτική επιστήμη, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Ούτως ώστε να υπάρχει μία ισορροπία, μία αντιστοιχία με τις κοινοβουλευτικές ομάδες που αποτελούν το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο ώστε να υπάρχει μια διαπραγμάτευση που να καταλήξει σε κάποια πρόταση, αντιπρόταση ότι είχε σε έκπληξη η κατάσταση που διαμορφώθηκε. Και ο Ζράμος, ο οποίος είπε εξ όμως της κυβέρνησης ότι πρόκειται να στηρίξει τον σημερινό πρόεδρο παρά το ότι ανήκει σε αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο. Ήταν επομένως αυτό μια έκπληξη. Τίποτα, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τίποτα δεν είναι απίθανο, λέει ο κύριος ε, Κασάδο. Η κυρία Ψολκόφσκα. Ε, το θέμα ήταν ε, του πώς θα προλάβουμε να συρρυκνώσουμε τις συνέπειες της κρίσης. Αυτό το, το, το πάλεψαν όλες τις δυνάμεις πριν τις εκλογές. Άρα εσείς ε, τι λέτε κύριε Επιτροπή, πώς θα έπρεπε να έχετε περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να μπορείτε να κάνετε κάτι σε τέτοιες καταστάσεις, Βάλστρομ. Το θέμα είναι τι θα γίνει στη συνθήκη της Λισαβόνας, εάν θα προχωρήσει η υπόθεση της συνθήκης και να αποδοθούν αυτές οι αρμοδιότητες, ούτως ώστε να μπορεί η Ευρώπη να κάνει αυτά τα οποία θέλει. Και το θέμα είναι ποιος θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μία φωνή που μιλά για την Ευρώπη στα διεθνή φόρα. Αυτό ήταν η υψίστη προτεραιότητα από τότε που αρχίσαμε να συζητάμε μετά τις οικονομικής κρίσης και νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα αντέδρασε η Επιτροπή Μπαρόσο που προσπάθησε να επισημάνει τι συμφέροντα διακυβεύει η Ευρώπη σε όλα αυτά. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει εν συνεργία, εν συνεργασία να αντιδράσουμε στην κρίση. Είναι θέμα το οποίο συνέχεια μας απασχολεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, γιατί έτσι κανείς κερδίζει σε νομιμότητα ως προς τους ψηφοφόρους αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αντιμετωπίσει, να χειριστεί τις κρίσεις και τα αυθεντικά, τα πραγματικά πολιτικά προβλήματα, τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Άρα Έχουμε τα μηνύματα, έχουμε τα διδάγματα από τη σημερινή μέρα. Προ πολιτικέ ομάδε και προ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μήνυμα είναι να μην φοβάστε την πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί αυτό το καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι. Επίσης, δίδαγμα προς τα κράτη-μέλη. Σιγουρέψτε το ότι η Ευρώπη είναι παρούσα στι συζητήσει στο ιστορικό του κράτου. Να μην συζητάτε μόνο τα εθνικά θέματα σε ευρωεκλογέ. Και δίδαγμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να συνεχίσει την συνεργασία. Να συνεχίσει το να εξηγεί τα θέματα καλύτερα. Αλλά το, το μήνυμα είναι να εκπροσωπούνται περισσότερο οι γυναίκες σε όλες τις θέσεις, σε όλα τα επίπεδα στο μέλλον. Uh, τα προβλήματα είναι ότι ο κόσμος και οι κυβερνήσεις ε, πρεσβεύουν ότι θέλουν περισσότερη Ευρώπη, μεγαλύτερη Ευρώπη με εξουσίες, αλλά δεν θέλουν να χωρίσουν την εξουσία αυτή στα θεσμικά όργανα γιατί θα τη χάσουν οι ίδιοι. Κύριε Πέρισιτς, εσείς τι πιστεύετε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι έτοιμοι να δώσουν μεγαλύτερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ευρωπαίοι, οι λαοί δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να κατανοήσουν τα θέματα αυτά και να τα συζητήσουν. Αυτά που ξέρουν οι πολίτες είναι τα όσα τους λένε οι κυβερνήσεις εμπολής. Και οι κυβερνήσεις λένε ότι οι Βρυξέλλες είναι κακές. Εκτός ε, όταν ισχυρίζονται ότι εκείνοι πέτυχαν μεγάλες νίκες στις Βρυξέλλες και αυτό οφείλεται στις κυβερνήσεις, όχι στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις, οι περισσότερες έτσι, δεν θέλουν να χωρίσουν περισσότερες εξουσίες στα θεσμικά όργανα γιατί θέλουν να τα κρατάνε στα χέρια τους αυτά. Είναι διατεθειμένες να το κάνουν μόνο εφόσον υπάρχει σαφής απόδειξη ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος και δεν γίνεται διαφορετικά. Ανέκαθεν ήταν αυτή η κατάσταση. Εδώ όμως έρχεται ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Επιτροπής και Κοινοβουλίου να το εξηγήσουν. Λυπάμαι ε, την Επίτροπο Βάλστρομ, αλλά ε, ήταν ε, εντυπωσιακά απούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κρίση αυτή. Μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγαίνει ασπροπρόσωπη από την κρίση. Το Κοινοβούλιο ήταν παραμονές εκλογών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν το ασχημόπαπο εκεί που δεν τολμούσε να αρθρώσει λόγο και η μόνη που αντέδρασε ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι δε κυβερνήσει μας ε, είπαν ότι μπορούν να ε, αντιμετωπίσουν την κρίση με συντονισμό. Μα είναι σαφέ ότι δεν μπορούν. Αυτό όμω δεν το εξήγησαν ποτέ στην κοινή γνώμη. Συμφωνώ με τον Μάριο Σέπη η προεκλογική εξαρτία έγινε από τις κυβερνήσεις με εθνικά κριτήρια. Αλλά η άλλη μεγάλη αποτυχία είναι τα λεγόμενα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ποια, τα ανύπαρκτα. Είχαν μια θαυμάσια ευκαιρία να ε, κάνουν πολιτικό ζήτημα το θέμα του διορισμού του επομένου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απέτυχαν σε αυτό. Δεν υφίστανται ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Καλά υπάρχουν ε, μόνο όταν πρόκειται να μοιράσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τις θέσεις και τα λάθη. Αλλά χάραν αυτή την ευκαιρία, δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλο. Και πέρα από τη χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές θα δούμε και ένα άλλο αποτέλεσμα που είναι η αύξηση των ακραίων και ε, λαϊκιστικών κομμάτων δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι ένα ε, σημείο πάρα πολύ ανησυχητικό. Όχι μόνο για την Ευρώπη την ίδια, αλλά και για τη δημοκρατία στις χώρες μας, όλες τις χώρες. Από ό,τι φαίνεται από τα πρώτα αποτελέσματα, τα ακροδεξιά και εθνικιστικά κόμματα τα πηγαίνουν πολύ καλά. Κύριε καθηγητά, Σύνοτο, αυτό το θεωρείτε πλέον τάση εδρεωμένη στην Ευρώπη και θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι σε περίοδους κρίσεων έχουμε περισσότερο εθνικισμό. Κοιτάξτε, το πρώτο μεγάλο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό ήταν κάτι σχετικά εύκολο να γίνει. Διότι Βεβαίω χρειαζόταν μεγάλη πρωτοβουλία και νόμοι, και, αλλά αυτό που χρειαζόταν ε, ήταν μια πολιτική βούληση και συμφωνία ότι ήταν απαραίτητο. Αλλά έχουμε και τώρα ένα φάσμα πολιτικών θεμάτων που είναι πολύ πιο δύσκολα ορισμένα. Θέματα, για παράδειγμα, μετανάστευση ή πολυφωνία και όλα αυτά. Ε, οι πολίτες τα θεωρούν πολύ πιο απτά από κάποια άλλα. Και σε περίοδους κρίσεως όπως αυτή που διανύουμε ε, μπορεί ε, αντίστοιχα να υποστηρίσουν ακραία κόμματα. Η μόνη άμυνα εκεί είναι να είναι πολύ ε, γερά τα επιχειρήματα και η συζήτηση στα μεγάλα κόμματα και είναι πραγματικά αδύναμα τα μεγάλα κόμματα στην ευρωπαϊκή τους διάσταση. Αλλά είναι δύσκολο να διαδεί κανείς πώς θα το ξεπεράσουμε. Είναι ε, μια διαδικασία που χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη πολιτικοποίηση της συζήτησης. Δεν εννοώ τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, αλλά τη δημόσια και συμμετοχή με άλλα θεσμικά όργανα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια διαδικασία συνασπισμών ε, μεταξύ πολιτικών κομμάτων αλλά και συμμαχιών μεταξύ θεσμικών οργάνων. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση. Είναι ουσιαστικά ελάχιστες οι αλλαγές. Μέχρι και οι Δανείοι δηλαδή αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε γιατί είναι μηδαμινές οι αλλαγές. Δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση έτσι ο κόσμος και ούτε βλέπω και μεγάλες ορέξεις και, ε, για αλλαγή στο μέλλον. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες. Έχουν ζητήσει δύο ε, κύριοι το λόγο και ο κύριος Σέπη και ο κύριος Μπέριτσιτς. Ε, ε, μια που μιλούμε για ευρωπαϊκά κόμματα, ενδεχόμενα ευρωπαϊκά κόμματα, υπάρχει ένα κίνημα που γεννήθηκε ακριβώς στην Ιρλανδία με το φαινόμενο Λίμπερτας που τώρα επιχειρεί να προσλάβει πανευρωπαϊκές διαστάσεις, που δεν είναι ακριβώς υπέρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Οπότε Καλύτερα τα καταφέρνουν οι αντιευρωπαϊστές ε, στο να κάνουν ένα κοινό κίνημα παρά εκείνοι που είναι υπέρ τη Ευρώπης. Τι λέτε κύριε Σέπη. Ήθελα να πω ότι η δημιουργία της ενιαίας αγοράς ήταν θεμελιώδης χαρακτήρα, ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για να πραγματοποιηθεί. Αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι ακόμα που είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση την Ευρωπαϊκή Συντογματική Συνθήκη, νομίζω ότι μπορούμε να τη λέμε ακόμα έτσι και όχι η Συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί είναι σημαντική, γιατί αυτή η συνθήκη περιλαμβάνει στο εσωτερικό της μια σειρά από τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας δυναμικής διακυβέρνησης της Ευρώπης, μιας ευκυβερνησίας πολύ πιο προωθημένης, η οποία ξεκινάει από μια προεδρία της Ευρώπης με ένα πρόεδρο ο οποίος θα έχει μια θητεία 2-2,5 ετών ανανιώσιμη και επίσης με την ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν το υποτιμώ. Εκεί που έχει προβλήματα η συνθήκη αυτή είναι ότι είναι δυσανάγνωστη για τους πολίτες της Ευρώπης. Δεν την καταλαβαίνουν οι πολίτες. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ακόμα και αν είναι μονάχα ένα προσαρτημένο πρωτόκολλο, θα γίνει κατά την άποψή μου ένα σημαντικό στοιχείο τη. Ε, ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Επίσης η ευρωπαϊκή ταυτότητα, αυτό το μήνυμα που δίνει η Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης το πρόβλημα των ε, ξενοφόβων και των ε, ρατσιστικών κινημάτων, με τα οποία συνδέεται σε κάποιο βαθμό η Λιμπέρτα. Εγώ πάντως δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μια κρίσιμη μάζα η οποία μπορεί να αλλάξει τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τα κόμματα αυτά έχουν μια μεγαλύτερη πρόσβαση στην κοινή γνώμη και δημιουργούν το φόβο για τον άλλο, μια, ένα κλίμα φοβία, το οποίο δεν μπορεί να το επιτρέψει η Ευρώπη στον εαυτό τη. Η Ευρώπη δεν πρέπει να φοβάται του άλλου. Θα πρέπει να είναι αυτή η οποία δίνει το παράδειγμα στου άλλου. Και τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρο τη κοινή γνώμη αρχίζει να δέχεται μια τέτοια ξενοφοβική αντιμετώπιση θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο μια τέτοια θέση κοινωνίας των πολιτών. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε με την ευρωπαϊκή μέθοδο, με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Ο κύριος Πέριτσι για ένα ερώτημα εδώ. Είναι μια πάρα πολύ ευρύ... διαδεδομένη συνήθεια αυτό το να θεωρηθείτε ότι ό,τι έγινε είναι εύκολο, αλλά αυτό το οποίο έρχεται την επαύριο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο. Όταν υπεγράφει η συνθήκη της Ρώμης, πολλοί είπαν ότι η Τελωνική Ένωση ποτέ δεν θα λάβει σάρκα και οστά γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Και πάρα πολλοί είπαν μετά ότι η ενιαία αγορά είναι κάτι το αδύνατο να επιτευχθεί. Και πολλοί είπαν δεν θα υπάρξει ποτέ Ευρώπη. Και τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι το αύριο είναι δύσκολο. Κλασικό αυτό, κλασικό αυτό για την Ευρώπη. Εγώ νομίζω, λέει ο κύριος Συνότο, ότι αυτό είναι κάτι ε, το οποίο ή αποτελεί μία πολιτική διαδικασία. Αποτελεί ε, την, την πρόσδοση ενός χαρακτήρα πολιτικού. Αυτό αφορά την ολοκλήρωση. Όσο προχωράει η ολοκλήρωση, γίνεται όλο ένα και πιο φορτισμένη πολιτικά και αυτό θα πρέπει να διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα. Έχετε δίκιο. Εάν όμως αυτό το οποίο είχαμε επί της τραπέζης αφορούσε την εγκαθίδρυση ενός ομοσπονδιακού, ομοσπόνδου ευρωπαϊκού κράτους, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εάν έρχεστε και μας λέτε ότι το κοινό νόμισμα δεν είναι πολιτικό, πολύ πολιτικό θέμα, ε, φυσικά και είναι και το καταφέραμε και πρόκειται για σημαντική επιτυχία. Να, ως παράδειγμα κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί απολύτως αναγκαίο. Στη τελευταία συνάντηση των 20 πιο προηγμένων χωρών στο Λονδίνο του G20 υπήρχαν δύο Αμερικανοί, ένας Κινέζος και δέκα Ευρωπαίοι. Αυτό μου φαίνεται γκροτέσκο. Ε, ε, παράλογο, κα, κανείς δεν τους πήρε στα σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε τη συμμετοχή της Ευρώπης στη διαχείριση του παγκοσμίου συστήματος εάν έχουμε 10 Ευρωπαίους να κάθονται γύρω γύρω από το τραπέζι. Έλεγαν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης ότι σκοτωνόντουσαν για το ποιος θα πρωτομπεί σε αυτή την ε, συνάντηση. Θεωρούσαν ε, το ότι όσο πιο σημαντικό γίνεται το G20 τόσο συρρυκνώνεται το ειδικό βάρος της Ευρώπης την ώρα της εκπροσώπησης. Τι λέτε. Κύριε Βάλστρομ, οφείλω να σας πω ότι η μνήμη στην πολιτική είναι πάρα πολύ σύντομη. Βραχία. Βεβαίω και είστε ελεύθερο να λέτε ό,τι θέλετε για και φιλοδοξίε κλπ. όσον αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά το θεσμικό όργανο το οποίο σε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπεραμείνθηκε της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήμασταν οι πρώτοι και οι μόνοι οι οποίοι προσπαθήσαμε να υπάρχει και η οπτική γωνία της Ευρώπης σε αυτή την υπόθεση. Γιατί πρώτα πρώτα, όπως θυμάστε, μεγάλες χώρες αρνήθηκαν την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε διαφορετικές φάσεις όλες οι μεγάλες χώρες υιοθέτησαν προστατευτικά μέτρα και εκεί μπήκε στο παιχνίδι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδραμάτισε τον ρόλο τη. οπότε δεν μπορώ παρά να υπεραμεινθώ των δικών μας ενεργειών. Και γι' αυτό βεβαίως και στο G10 και στο G20 έχουμε τη θέση μας τόσο ώστε να μπορούμε να κάνουμε να ακουστεί η φωνή της Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για το μέλλον. Να μην είμαστε κοινικοί, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν επιτευχθεί τα οποία τα έχουμε κατακτήσει και θα πρέπει να γνωρίσουν κάποια συνέχεια, ούτω ώστε να διαμορφώσουμε κάποιο είδους πολιτικό θεμέλιο στην Ευρώπη. Είδατε. Φυσικά και όλα αυτά έχουν βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και παραπέρα, θα πρέπει να γίνουν πραγματικά πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, θα πρέπει και στην εσωτερική πολιτική ε, προβληματική να μπουν τα ευρωπαϊκά θέματα, θα πρέπει Επομένω, η, να, να, να, έχει τι ρίζε της η ευρωπαϊκή πολιτική στα εθνικά πολιτικά κόμματα. Ιδάλω, είναι αδύνατο να κινητοποιηθούν οι εθνικοί, οι, οι, οι ψηφοφόροι στα κράτη-μέλη. Μισό λεπτό, Χριστίνα. Θα σου δώσω το λόγο, αλλά πρώτα πρώτα θέλει το λόγο να μα πει δύο κουβέντε ο κύριο Κασάδο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πήγαινε στο G20 δεν συρρυκνώνει το ειδικό βάρο τη ε, Ευρώπη. Γιατί αυτό το οποίο θίγεται είναι το G8 από το G20. Ε, ε, γιατί μιλάμε για την διεθνή σκηνή. Είναι οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις συν η Ρωσία. Είναι οι αναδυόμενες χώρες, είναι οι χώρες οι λιγότερο ανεπτυγμένες και πρόκειται για μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα η οποία σχηματοποιείται από το G20 και βεβαίως η Ευρώπη πρέπει εκεί να πηγαίνει και να ακούγεται μία φωνή της έχουμε την αυξανόμενη σημασία της Κίνας αλλά και της Ευρώπης οπότε θα πρέπει και η Ευρώπη με μία φωνή να εκφράζεται σε αυτά τα φόρα. Κάτι το οποίο θα βοηθηθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όλοι οι φιλοευρωπαϊστές θέλουμε η διαδρομή αυτή να έχει ο τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα Τη διαδικασία αυτή τη παγκοσμιοποίηση, ούτω ώστε έτσι να σχηματοποιηθεί η νέα κατάσταση. Είναι αδύνατον αλλιώ να πηγαίνει στα διεθνή φόρα η Ευρώπη, εάν δεν πηγαίνει και να ακούγεται ενιαία η φωνή τη. Έχω κάποια στοιχεία τώρα, νομίζω ότι είναι η τελική συμμετοχή στις εκλογές που υπολογίζεται σε 43 περίπου τα 100. Είναι αυτό το οποίο περιμένατε εσείς, αυτό προβλέπατε σαν ποσοστό συμμετοχής. Οι πρώτες ε, αναφορές που είχαμε ήταν πάρα πολύ απεσιόδοξες και τα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει προβλέψεις πολύ χαμηλότερες από αυτό που βλέπουμε σήμερα σαν τελικά ποσοστά συμμετοχής. Περιμέναμε βέβαια ότι θα είχαμε μια ανάμεικτη εικόνα. Απλώς όμως αυτό μας δείχνει ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, να μάθουμε μάλλον από την κατάσταση των κρατών μελών θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πλησιάσουμε περισσότερο πολίτες. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω, κύριο Σίνετ, λέει, ότι δεν νομίζω ότι είναι απλώς ανάμεικτη εικόνα, είναι αρνητική εικόνα. Μα Αν σκεφτούμε πόση προσπάθεια έγινε, πόσο μεγαλύτερη ήταν η λειτουργία του συντονισμού μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχέδιά σας για μια εκλογική στρατηγική, όλα αυτά που έγιναν και όμως πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας τι είναι αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο αν ισχύουν τα στοιχεία αυτά της ε, <clears throat> συμμετοχής, βλέπουμε ότι κατά 3 ή 4% μειώθηκε πάλι η συμμετοχή. Και αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται και η δημοκρατική νομιμότητα του Κοινοβουλίου. Εάν πράγματι δεν μπορεί να πλησιάζει τους πολίτες και να συνδέονται οι πολίτες και οι χώρες μέλη με αυτά που γίνονται και συζητούνται στις Βρυξέλλες και το Στρισβούργο. Μα τι μπορείτε να περιμένετε, δεν είναι χαζή η εκλογής. Είχαμε μια εκστατεία η οποία ήταν καθαρά εθνικού χαρακτήρα, αποκλειστικά εθνική. Αλλά δεν ήταν για εθνικές εκλογές βέβαια. Ήταν ένα είδος δημοσκόπησης σε πραγματικό μέγεθος. <clears throat> και ο καθένας ψήφισε βάσει των πεπιθήσεών του για την εθνική πολιτική ζωή. Δεν υπήρχε ευρωπαϊκή διάσταση στις εκλογές αυτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί σε διάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο η συμμετοχή των εκλογέων ήταν κάτω από 50% και όμως είναι ένα από τα πιο νομιμοποιημένα κοινοβούλια στον κόσμο το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με 43% συμμετοχή των εκλογέων θέλει να ασκήσει τις, εξογε... εξουσίες που έχει, είναι πράγματι νομιμοποιημένο. Κανείς δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθεί για κάτι τέτοιο. Μπορεί την επόμενη φορά να έχουμε και μεγαλύτερη προσέλευση των εκλογέων, αν και όταν σημειώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό, ότι ο τρόπο για να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση είναι ακριβώ με το να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική συζήτηση και πολιτικοποίηση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Και υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό το οποίο λένε οι πολιτικολόγοι εκλογή δευτεροκλασάτη, δεύτερης κατηγορίας η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να αντιμετωπίσετε σαν κανονική εκλογική διαδικασία, ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μείωση της ε, προσέλευσης, αλλά είναι περιορισμένη. Εγώ νόμιζα θα ήταν μεγαλύτερη. Νομίζω ότι ο Ευρωπαίος ε, εκλογέας θα νόμιζε ότι περίπου τον κοροϊδεύουν κάτω σε αυτές τις συνθήκες γιατί του ζητάνε να εκλέξει ευρωβουλευτέ επί τη βάση τη εθνική προβληματική. Και νόμιζα ότι θα ήταν ακόμα μικρότερο ο αριθμό των Ευρωπαίων που θα πήγαινε να ψηφίσει, γιατί είναι σαν να του λες κάνε μια χάρη στο εθνικό μου κόμμα, ψήφισε με στην Ευρώπη. Αλλά τελικά ήμουν υπερβολικά απεσιόδοξος. Από την άλλη μεριά, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. <clears throat> γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερε εξουσίε. ελπίζω με τη συνθήκη τη Λισαβόνα θα γίνει αυτό. Έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν εξουσίες, αλλά πρέπει να ανταποκριθεί στι απαιτήσει των εκλογέων. Για μένα λοιπόν αυτή η σχέση εκλογέων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα. Εμεί λοιπόν θεωρούμε ότι αν τέθει σε εφαρμογή η συνθήκη τη Λισαβόνα, αυτό θα ενισχύσει ιδιαίτερα τη συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ακόμα και μέσα από τα θεσμικά, τα παραδοσιακά θεσμικά κανάλια να συμμετέχουν λοιπόν η κοινωνία των πολιτών στα δημόσια πράγματα. Το να υπάρχουν λοιπόν μη κυβερνητικέ οργανώσει ή ενώσει των πολιτών που συμμετέχουν, αυτό θα δώσει μια νέα νομιμοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είχαμε συντάξει ένα πρόγραμμα στο οποίο είχαμε 22 αν θέλετε θέματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Και μέσα σε αυτά τα, αν θέλετε, τα πλαίσια μέσα στα οποία θέταμε τα διάφορα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε καταθέσει 87 συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτό είναι δικό μας ε, εγχείρημα, είναι δική μας αρμοδιότητα γιατί σαν Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή πρέπει να βοηθήσουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο των Υπουργών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν καταφέρουμε να αναπτύξουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με την Κομισιόν, την τρέχουσα Κομισιόν, μια συζήτηση για να υπάρξει συνεργασία για τα θέματα αυτά, αυτό θα δώσει μια ανανομιμοποίηση στο Κοινοβούλιο, διότι θα έχει δώσει πραγματική απάντηση στα προβλήματα τη Ευρώπη. Αν ε, κάτσουμε και λάβουμε υπόψη αυτό το οποίο είπατε, θα πρέπει να κάνουμε αναχώρα ανάλυση αυτών των μεταβλητών για να δούμε ακριβώ τι γίνεται με την εσωτερική πολιτική. Δύο λεφτάκια μας μένουν, οπότε η σκητάλη τώρα στην Χριστίνα. Για πέστε μας για το σύμφωνο σταθερότητας. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει, κύριε τις επαναλαμβάνω, θέλω να σας ρωτήσω για το σύμφωνο σταθερότητας. Ναι, Πέρεσιτς. Ναι, υπό την σημερινή συγκυρία με αυτή την ε, έντονη ύφεση θα πρέπει να έχουμε ως οροφή ελλείμματο το 3% όμως αυτό πώς είναι δυνατόν αφού από την άλλη μεριά έχουμε αρνητική ανάπτυξη και από την άλλη ε, μεριά έχουμε τις πιέσεις από την κρίση. Επομένως, το σύμφωνο σταθερότητας μπορούμε να πούμε ότι τώρα ε, είναι κάτι το απειρχιωμένο. Παρακαλούμε πολύ σύντομη συγκεκριμένη απάντηση. Όχι, όχι. Η κυρία Μέρκελ το έθεσε πάρα πολύ καλά όταν είπε χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι η πιο δύσκολη στιγμή θα είναι όταν ανακάμψουμε από την κρίση, διότι προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Διότι θα πρέπει να ρίχνουμε ρευστό στην αγορά προς το παρόν. Όταν όμως σταματήσει η κρίση, τότε θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην ορθολογιστική διαχείριση των δημοσιονομικών, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να γίνει. Χουάν Πέδρο. Ήρθε η σωστή στιγμή που νομίζω ότι και ο κύριος Κασάδο θα είχε πολλά να μας πει σε σχέση αλλά και ο κύριος Σύνοτο όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο ήρθε η ώρα. Είναι 9.30 Είδατε πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα. Ε, τι να κάνω. Συμπαθάτε μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλοι μαζί μας και θα τα πούμε στην επόμενη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε.